Αν θέλετε καθίστε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Το δε πρώτο είναι η μερίσια διάταξη, την οποία σας διαβιβάσαμε Δευτέρα απόγευμα. Αν δεν έχετε, ορίστε, ο κ. ομαρζή. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Υπενθυμίζω πρώτα το άρθρο 130, παράγραφος 5 του κανονισμού, σχετικά με τις γραπτές ερωτήσεις. Τι λέει το άρθρο αυτό? Εάν ερώτηση δεν απαντηθεί μέσα σε προθεσμία τριών εβδομάδων, πρόκειται για κατά προτεραιότητα ερωτήσεις ή έξι εβδομάδες για μη κατά προτεραιότητα ερωτήσεις, οι οποίες εβδομάδες μετρούν από την αποστολή της, μπορεί μετά από αίτηση του ερωτώντος να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδριάσεως της Αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Στις 18 λοιπόν Δεκεμβρίου απίφθηνα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ερώτηση κατά προτεραιότητα, για την ανεξαρτησία από το σύστημα, το σύστημα τους μάλλον ε, καπνού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εχνητασιμότητας. Δεν έχω λάβει απάντηση μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο κανονισμός. Και δικαιώσατε το αίτημά μου, δηλαδή να εγγραφεί στην ημερησία διάταξη της Επιτροπής μας η ερώτηση αυτή. Και πράγματι στις 20 Φεβρουαρίου την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, η ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας περιλάμβανε την ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ερώτηση επαναλαμβάνω που δεν είχε απαντηθεί. Και σας ομολογώ ότι είμαι ιδιαίτερα έκπληκτος που είδα ότι την Δευτέρα αποσύρθηκε η ερώτησή μου από την ημερήσια διάταξη. Είμαστε κοινοβουλευτικοί εδώ, έχουμε κάποια δικαιώματα που τα περιλαμβάνει ο κανονισμός. Και για την ίδια την αξιοπιστία του θεσμού μας, του Κοινοβουλίου, αλλά και λόγω σεβασμού απέναντι στους κοινοβουλευτικούς, είναι ευθύνη σας ως Προέδρου να εφαρμόσετε τον κανονισμό. Για τον λόγο αυτό διερωτώ με. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν να αποσύρετε την ερώτησή μου από την ημερήσια διάταξη. Και οφείλω να διαπιστώσω ότι όταν πρόκειται για την βιομηχανία καπνού, πάντοτε βλέπουμε το ίδιο. Δηλαδή πολλές περιπλοκές. Ήθελα λοιπόν να ερωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελειώνω με αυτά τα λόγια σχετικά με την απόφασή της έγκρισης του Οκτωβρίου 2018 για τον κατάλογο αποθηκών που είχε δώσει η βιομηχανία καπνού και τον Δεκέμβριο του 2018 επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να κάνει προκήρυξη διαγωνισμού και έχει περιλάβει όλους τους ιστορικούς παράγοντες της βιομηχανίας καπνού. Την τελευταία, ε, την περσινή χρονιά, είχα θέσει θέματα του παράλληλου εμπορίου προϊόντων καπνού. Πρόκειται για φάκελο σημαντικό. Από τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει σε ισχύ το σχετικό πρωτόκολλο και εμείς έχουμε υποχρέωση να θέσουμε ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του συνόλου του κανονισμού αυτού που προβλέπει το πρωτόκολλο. Άρα υπήρχε ένα θέμα, το οποίο θέμα έπρεπε να περιλαμβάνεται στη μέση διάταξη του σημερινού πρωινού. Δεν θα σας ζητήσω να περιλάβετε την ερώτηση αυτή μέσω ψηφοφορίας στη σημερινή μερίσια διάταξη, διότι ούτως ή άλλως αυτά θα αποτελούσε καταστρατήγηση του κανονισμού. Είμαι κοινοβουλευτικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μου απήντησε, δεν μου απήντησε ευθέω. Θεωρώ ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι σήμερα παρούσα για να μπορέσω να την ερωτήσω. Σα ευχαριστώ. Η πρόεδρο Βαλέαν, ευχαριστώ κύριο Μαρζή. Έχετε βέβαια Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι η, η Κομισιόν θα έπρεπε να έχει απαντήσει στην ερώτησή σας. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδωσε κανένα μήνυμα ότι θα απαντήσει. Στο μεταξύ έχουν στείλει την ε, απάντηση στα αγγλικά και σας την έχουμε διαβιβάσει. Και στο τέλος της εβδομάδος θα έχετε και το γαλλικό κείμενο της απάντησης. Γι' αυτό το λόγο η γραμματεία πρότεινε να αποσυρθεί το θέμα από την ημερησία διάταξη, γιατί στο μεταξύ έχει έλθει η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν θέλετε να διεξαρθεί συζήτηση στη σημερινή ημερήσια διάταξη, γιατί θέσατε κάποια ερωτήματα, τότε μέσω του συντονιστού σας να το προτείνετε. Και θα μπορέσουμε να περιλάβουμε, να αποδεχθούμε το αίτημά σας, εφόσον συμφωνήσουν και άλλες πολιτικές ομάδες, ώστε να περιληφθεί τέτοιο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Για το συγκεκριμένο θέμα της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προφανώς ήρθε η απάντηση, βέβαια μόνο στα αγγλικά. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τι άλλο να σας πω. Θέλετε να το προχωρήσετε το θέμα αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν ζητάτε σήμερα να μπει στην ημερήσια διάταξη. Μιλήστε λοιπόν στο συντονιστή σα. να το συζητήσουν μετά οι συντονιστέ μεταξύ των, ώστε να μπει σε μια μελλοντική μερίσια διάταξη. Δεν σα αρέσει αυτό. Αλλά παρακαλώ σύντομα, λάβετε το λόγο, αλλά σύντομα, γιατί έχουμε και συζήτηση να κάνουμε. Ο Μαρζέ. Θέλω να πω μόνο ότι όταν κανεί είναι βουλευτή, τα κάποια προνόμια που διαθέτουμε προέρχονται από την άμεση και αυστηρή εφαρμογή του δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να απαντά ευθέω και άμεσα μέσα σε τρει ή έξι εβδομάδε με άμεση απάντηση στον βουλευτή. Κάτι το οποίο δεν έπραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν προκειμένου. Έχω λοιπόν το δικαίωμα να ζητήσω, χωρί να περάσω από τον συντονιστή, να εγγραφεί το θέμα μου στην ημερήσια διάταξη. Και εσεί συνενέσατε. Εν τω μεταξύ αποφασίστηκε και είπατε μάλιστα ότι ήταν ε, το προσωπικό τη γραμματεία που αποφάσισε να αποσύρει το θέμα από την ημερήσια διάταξη. Αυτό που ζητώ δεν είναι απόφαση των συντονιστών. Ζητώ την εφαρμογή του κανονισμού. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβα απάντηση ευθέω σε μένα. Μπορούν να μου απαντήσουν σε όποια γλώσσα θέλουν, αλλά δεν έχω λάβει άμεση απάντηση προ εμένα προσωπικά. Άρα, κανονικά θα έπρεπε σήμερα να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απάντηση τη Πρόεδρου Βαλαιάν. Α το σταματήσουμε εδώ κύριε Μαρζέ. Σημείωσα τα όσα είπατε. Έχετε λάβει την απάντηση. Ασφαλώς δεν ήταν τέλεια η διαδικασία. Η, η μερίσια διάταξη είχε διαβιβαστεί στους συντονιστές με την τροποποίηση αυτή. Δεν έλαβα καμιά ενστασία από τον δικό σας συντονιστή. Τι άλλο να σας πω. Έχετε την απάντηση στο μεταξύ. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Αλλά νομίζω... Όχι, όχι λέει ο κύριο Σόμοζη αλλά χωρίς μικρόφωνο, κατά τα λοιπά. Άρα, δεν υπάρχει πρόταση τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης. Εγκρίνεται λοιπόν η ατελής αυτή η ημερήσια διάταξη σήμερα και έχω και κάποιες ανακοινώσεις, συνεχίζει η πρόεδρος Βαλιάν, για το Στρασβούργο, στις 14 Μαρτίου, δηλαδή 5η, 9 το πρωί. Σύντομη συνάντηση της Επιτροπής ΕΝΒΗ, γιατί θα έχουμε κάποιες αποφάσεις σχετικά με ψηφοφορίες που θα πρέπει να γίνουν με επίγοντα τρόπο. Θα σας διανεμηθεί έγκαιρα σχέδιο της ημερήσιας διάταξης για τη συνάντηση αυτή στις 21 Τρίτου απόγευμα η οποία είναι ακόμα σε ρεζέρβα. Έχουμε, ήταν μάλλον τώρα, έχουμε ακυρώσει τη συνάντηση αυτή. το απόγευμα. Το πρωί όμως θα γίνει συνεδρίαση. Σας προσκαλώ όλες και όλους, μετά θα σας προσκαλέσω δηλαδή, σε κοκτέιλ της ε, Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος για να ε, εορτάσουμε την ολοκλήρωση των εργασιών μας και τα λοιπά. Και στις 27 Μαρτίου, στο τέλος τη απογευματινής συνεδρίας που θα γίνει στο Στρασβούργο, θεώρησα σωστό να προσκαλέσουμε και τα πρόσωπα που έχουν συνεργαστεί μαζί μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίω όλα τα μέλη της ΕΝΒΗ. Σας παρακαλώ σημειώστε το στα ημερολογιά σας. Και αυτές ήταν οι ανακοινώσει μου. Έχουμε και τα πρακτικά. Τα πρακτικά της 21ης, 22ης και 29ης Ιανουαρίου. Εάν λοιπόν δεν υπάρξουν σχόλια θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Τώρα θα προχωρήσουμε σε ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για τα συστήματα μέτρησης εκπομπών αυτοκινήτων. Ε, παρόν είναι ο κύριος Τζάρεμπ, πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. και συντάκτης της έκθεσης που θα μας παρουσιάσει παρουσίασε μάλλον το briefing paper του ελεγκτικού συνεδρίου για την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο λεγόμενο Dieselgate. Επειδή εμείς έχουμε προωθήσει τη σχετική νομοθεσία, αναμένουμε με ενδιαφέρον την παρουσίαση του κυρίου Τζάρεμπ. Έχουμε... Έχετε το λόγο, κύριε Τζάρεμπ. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το έγγραφό μας για το λεγόμενο Dieselgate. Πρώτα, είχαμε ειδική έκθεση για την ατμοσφαιρική ρήπανση που είπαμε ότι είναι ο μεγαλύτερο κίνδυνος για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ατμοσφαιρική ρήπανση οδηγεί σε 400.000 πρόωρου θανάτου κάθε χρόνο και σε δισεκατομμύρια ε, κόστος υγείας. Και 40% και ένα 11% των σωματιδίων προέρχονται από τι εκπομπέ αερίων των αυτοκινήτων. Υπάρχουν συστήματα ελέγχου στο ε, επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτά απέτυχαν. Ενώ έχουν μειωθεί ε, οι ανώτατες τιμέ 200 από το 2000, οι ε, εκπομπέ αζότου έχουν συνεχιστεί ωστόσο. Το ελεγχτικό συνέδριο έλαβε έτοιμα από τη διάσκεψη Προέδρων Πολιτικών Ομάδων να κάνει έναν έλεγχο για τα συστήματα αυτά. Αποφασίσαμε εμείς να σας δώσουμε ωστόσο καλύτερα ένα briefing paper. Γιατί το κάναμε αυτό. Πρώτα, διότι η Επιτροπή σας έκανε μια θαυμάσια δουλειά για την εξέταση των σχετικών συστημάτων. Δεν θελήσαμε λοιπόν να επικαλύψουμε την εργασία σας. Δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει, λάβει, έχει αναλάβει δράσεις προτείνοντας νέα νομοθεσία απαντώντας στο εμείς, δηλαδή στα απορίσματα της, Επιτροπής, της Ειδικής Επιτροπής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο επίπεδο του ευρωπαϊκό και στο επίπεδο των χωρών μελών. Άρα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα audit, και επίση θελήσαμε να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκθεση πριν από τι ευρωεκλογέ, ώστε να μπορέσετε να δείτε τι έγινε μετά από την δημοσίευση της έκθεσης με τα πορίσματα της Επιτροπής ΕΜΗΣ. Το έγγραφο μας, ενημερωτικό έγγραφο δηλαδή, τονίζει τις αλλαγές που ενδέχεται να ε, επηρεάσουν την πατρισματική εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων. Και αυτό δεν περιλαμβάνουμε συστάσεις, αλλά αναφερόμαστε στις προκλήσεις για να βρεθεί ένας τρόπος να λυθούν. Αν δείτε τώρα τη θετική πλευρά του τι συνέβη ως ανταπόκριση δηλαδή στο σκάνδαλο Dieselgate. Το ίδιο το σκάνδαλο επιτάχυνε τις νομοθετικές ε, τροποποιήσεις για τους ελέγχους καυσαερίων με ενδυνάμωση των ε, αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να επανεξετάζει και να ελέγχει το έργο των εθνικών αρχών που ε, αναφέρονται στους ελέγχους εκπομπών, στην, ε, στις εγκρίσεις τύπων κλπ. Και νέα εργαστηριακά τεστ, το ε, παγκόσμιο εναρμονισμένο, εναρμονισμένη διαδικασία ελέγχου ελαφρών οχημάτων και αυτά είναι υποχρεωτικά τώρα για τις χώρες μέλη τα δηλαδή, δε ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη θα πρέπει να κάνουν επίσης ε, δοκιμασίες για εκπομπές. Εμείς βρήκαμε ότι υπάρχουν σημαντικά ωφελήματα από τα συστήματα αυτά RDA, RDE, διότι μειώθηκαν οι εκπομπές στην οδική κυκλοφορία από 800 σε 450 ε, μικρογραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Για τους, για τους κινητήρες που ε, είναι εξοπλισμένοι με συστήματα D6 με χρησιμοποίηση καταλυτών και ούτω καθεξής. Από την άλλη μεριά σημειώνουμε επίσης ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο το όφελος εάν το αρχικό όριο των 128 μικρογραμμαρίων ανά χιλιόμετρο είχε εγκριθεί αντί για το 168 μικρογραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Στο ενημερωτικό μας έγγραφο δεν περιλαμβάνουμε στοιχεία για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διότι εμείς εγκρίναμε τον ημερωτικό μα έγγραφο πριν εκδοθεί αυτή η απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολιτική η απόφαση για το πώ θα τροποποιηθεί η νομοθεσία στο προσεχέ μέλλον. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμεί είναι να σα ενημερώσουμε ότι βρήκαμε κάποια επιστημονική βάση σε επιχειρήματα και σε ό,τι αφορά τις αλλαγές, εμείς τονίζουμε ότι οι αλλαγές αυτές και ε, πρέπει να γίνουν στην νομοθεσία για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Θα βρουν οι κατασκευαστές νέες ευελιξίες και υπάρχει ο κίνδυνος ότι θα ε, βελτιστοποιήσουν τα οχήματα για το τεστ έντι και επομένως θα παραμείνουν υψηλές οι εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου. Η αποτελεσματικότητα τώρα των ελέγχων της αγοράς θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή που θα κάνουν οι χώρες μέλη. Και τα βασικά θέματα εδώ είναι ε, η ποσότητα των ελέγχων και η ανεξαρτησία των ελεγκτικών αρχών. Διότι μόνο σε δύο περιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι έλεγχοι, οι έλεγχοι αυτοί γίνονται από ανεξάρτητες ε, αρχές όπως οι ΗΠΑ. Και επίσης τονίζουμε ότι ε, το νέα, τα νέα τεστ από, ανεξάρτητες, ε, από ανεξάρτητα τρίτα μέρη ε, κινδυνεύουν να είναι πολύ περιορισμένα διότι είναι πολύ ψηλό το κόστος. Τώρα, υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται από τις πρόσφατες νομοθετικές δράσεις. Θα θέλαμε να τονίσουμε ιδίω ότι ίσως χρειαστούν πολλά χρόνια για να βελτιωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στα αστικά κέντρα λόγω των πολλών ε, των ε, πολυάριθμων αυτοκινήτων που προκαλούν υψηλή ε, ρήπανση, ενώ θα αρχίσουν να αποδίδουν τα μέτρα αυτά σε λίγα χρόνια. Πάνω από 10 εκατομμύρια οχήματα διαφόρων τύπων έχουν αποσυρθεί. Όμως, τα περιορισμένα διαδεμένα που διαθέτουμε δείχνουν ότι η μείωση των εκπομπών οξυδίων του αζώτου είναι πολύ μικρή. Το δε πλαίσιο για τις νέες εγκρίσεις τύπων εξαρτάται και από τις εγκρίσεις τύπων για τα νέα μοντέλα, αλλά αυτό δεν έχει επιτύχει στο παρελθόν. Θέλω επίσης να αναφέρω ότι ένα από τα σημαντικά θέματα είναι και ε, ότι ε, χειραγωγούν τα διάφορα συστήματα των ε, ε οχημάτων, των εκπομπών δηλαδή. Μέχρι τώρα αυτά εμπίπτουν στο εθνικό δίκαιο των χωρών μελών αλλά διαπιστώνεται μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων, αλλά πολλές χώρες μέλη δεν κάνουν περιοδικές, περιοδικούς ελέγχους εάν έχουν όντως αφαιρεθεί τα φίλτρα, κάτι το οποίο οδηγεί σε δεκαπλάσιους ή και ε, εικοσαπλάσια ποσά ε, εκπομπών. Αυτά είναι σύντομα τα ε, πορίσματά μας και αναμένω βεβαίω ευχαριστώ τις ερωτήσει σα για να τι απαντήσω. Well, Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, τώρα είναι η σειρά σας. Ποιος θέλει να μιλήσει για να συλλέξουμε παρατηρήσεις και ερωτήσεις για να επανέλθουμε στο ηλεκτρικό συνεδρίο για απαντήσεις. Παρακαλώ, κύριος ε, Γκερμπράντι. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, με εκπλήσουμε που είμαι ο πρώτος, αλλά θα ξεκινήσω ευχαριστώντας το ελεγκτικό συνέδριο για την μελέτη αυτή. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και τα πορίσματα της ευθυγραμμίζονται απολύτως με την Επιτροπή έρευνη, με την Επιτροπή μας εδώ και με την συζήτηση που είχαμε την περισμένη εβδομάδα με την Επιτρόπο Μπιανκόφσκα στην ΕΝΒΗ πολλά μπορεί να ρωτήσει κανείς σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες της έκθεσης. Ίσως βέβαια αυτό να μην είναι το κατάλληλο βήμα για κάτι τέτοιο. Με ικανοποιεί η επίκριση που κάνετε στους ε, παράγοντες συμμόρφωση και τεχνικός. Είναι ενδιαφέρον να βλέπει κανείς ένα υπεύθυνο φορέα όπως είναι το ελεγκτικό συνέδριο να επικρίνει την προσέγγιση αυτή. Ίσως να σας είναι δύσκολο να σχολιάσετε, αλλά εφόσον επέλεξε η Κομισιόν να προσφύγει κατά της τοποθέτησης του συνεδρίου, είναι κάτι που εκπλήσει. Τώρα, σχετικά με την ε, παρακολούθηση της αγοράς ε, και της αδυναμίας τα κενά του υφισταμένου στήματος όλα εξαρτώνται από την υλοποίηση από τα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια δυναμία δομική, θα έλεγε κανείς, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εγώ καλώ για μια υπηρεσία παρακολούθησης, επιτήρησης εδώ και χρόνια, ίσως κάποια μέρα να τα καταφέρουμε, αλλά στο μεταξύ υπάρχει μια λύση που θα μπορούσε να βοηθηθεί από το ελεκτικό συνέδριο. Γνωρίζω ότι έχετε πολύ καλές ε, σχέσεις με τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια, για τα οποία θα μπορούσε να είναι ε, αυτό το θέμα πολύ ενδιαφέρον, καθότι μιλούμε για κακή εφαρμογή της νομοθεσίας. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσατε να συζητήσετε με τους εθνικούς σας ομολόγους, ώστε να έχουμε δηλαδή εθνικές συστάσεις και ώστε τα ε, κρατικά εθνικά συστήματα να βελτιωθούν ουσιαστικά. Το άλλο που θέλω να αναφέρω είναι οι ελλείψεις που έχουμε σε επίπεδο λογισμικού και επικαιροποίηση. Συχνά βλέπουμε ότι δεν έχουμε επικαιροποίηση εξοπλισμού, αλλά τεχνικού εξοπλισμού, αλλά μόνο σε επίπεδο ηλεκτρονικού συστήματος, λογισμικού. Εσείς πώς θα θεωρούσατε ότι θα μπορούσε να επιβληθεί στην αυτοκινητοβιομηχανία να προχωρήσει σε επικαιροποίηση του τεχνικού της εξοπλισμού, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε στα αστικά μας κέντρα να γλιτώσουμε από όλες αυτές τις παράνομες εκπομπές εκατομμυρίων οχημάτων. Αυτά ήθελα να παρατηρήσω σήμερα και ευχαριστώ και πάλι το Ελεκτικό Συνέδριο για την εισήγησή του Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε. Άλλα μέλη λέει η πρόεδρος. Η κυρία Άβη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ ζήτησα το λόγο γιατί ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την παρουσίαση αυτή που είναι σημαντική. Η μελέτη αυτή ήταν σημαντικό επίσης να παρουσιαστεί δημόσια στην Επιτροπή αυτή και ώστε να διαχυθεί στο μέτρο δυνατού του περιεχόμενό της διότι υπογραμμίζει τα μεγάλα κενά και τις μεγάλες ελλείψεις που είχε σημειώσει το Κοινοβούλιο και τα κρατημέλη στα πλαίσια του σκανδάλου Dieselgate και όχι Volkswagen όπως είπα εκ παραδρομής. Ο συνάδελφος ήδη αναφέρθηκε σημαντικά σημεία αλλά ήθελα να επανέλθω στα στις αναδρομικές επικαιροποιήσει, τα retrofit όπως λέμε, στον εξοπλισμό των οχημάτων, διότι στο 64 σημείο της μελέτης σας αναφέρεστε ρητά στο ότι μπορούν αυτά τα retrofit να είναι εναλλακτική λύση απέναντι στην αναβάθμιση του λογισμικού. Αλλά κατά την άποψή σας Ποιε είναι οι απτές προτάσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει σε επίπεδο νοσιακό ώστε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση, διότι αυτό που είδαμε ήταν μια κατακαιρματισμένη ανταπόκριση και έλλειψη αρμονίας και σύμπνοιας μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτές οι επικαιροποιήσεις είτε δεν εγκρίνονται, δεν υιοθετούνται, είτε γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και πολύ περιορισμένα σε επίπεδο τεχνικού φυσικού εξοπλισμού. Τι λοιπόν πρέπει να γίνει ώστε αυτές οι βελτιώσεις, οι επικαιροποίησεις να λάβουν χώρα. Και κατά πόσον βρίσκεται και μία απόκληση, ε, έντονη απόκληση ανάμεσα στα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ και στα όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και η Volkswagen υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει τα οχήματα με αυτές τις επικαιροποιήσεις του τεχνικού, της, τεχνικού τους εξοπλισμού και επομένω βλέπω μια διάκριση μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών πολιτών λέει η ομιλήτρια και πιστεύω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κρατη θα πρέπει να, είναι, να έχουν περισσότερα κίνητρα προς, ώστε να αναλάβουν δράση. Και έκανα αυτήν την ε, ερώτηση στην Επίτροπο Μπιανκόφσκα την περασμένη εβδομάδα χωρίς να λάβω καμία απάντηση. Ήθελα να την επαναλάβω. Δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να δώσετε μια όθηση σχετικά με τη συμφωνία την πρόσφατη μεταξύ της Volkswagen και της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εγώ θα δοκιμάσω τώρα να αναφερθώ, εσείς αν μπορείτε θα το σχολιάσετε. Σχετικά με τη συμφωνία αυτή λοιπόν, η οποία αφορούσε σε 400 εκατομμύρια που δόθηκαν ως δάνειο στη Volkswagen τα προηγούμενα χρόνια και οι οποίοι πόροι δεν χρησιμοποιήθηκαν για την ε, μείωση των εκπομπών και έφτασε σε μια συμφωνία με την ΕΤΕ ε, σε διάφορα επίπεδα περιβαλλοντικού πιλωτικών έργων με δέσμευση επί 18 μήνες και σε ύψος 13 εκατομμυρίων. Τώρα, εγώ δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορείτε να σχολιάσετε, αλλά ε, εν πάση περιπτώσει δεν παρατηρείτε, δεν έχετε κάποια απορία, για να το πω έτσι, ως ελεκτικό συνέδριο σχετικά με τη συμφωνία αυτή. Δεν παρατηρείτε κάποια απόκληση, κάποιο σφάλμα. Σα ευχαριστώ κάποιο άλλο, Η Κομισιόν μήπω, Θα ήθελε το λόγο. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μητιοσύνη ονομάζομαι από την μονάδα αυτοκίνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ σύντομα θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, διότι ετέθη ξανά. λόγια για την αναβάθμιση λογισμικού σε σχέση με την αναβάθμιση του υλικού. Αυτή τη στιγμή ισχύει ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών η απόφαση για τον τύπο της διόρθωσης που είναι πιο κατάλληλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει για το αν, θα, ε, αν είναι πιο κατάλληλο υλικό ή λογισμικό για την ε, αναβάθμιση αυτή στην μετασκευή των οχημάτων. Να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να ε, γίνει μετασκευή με υλικό. Είναι ένα project εκατομμυρίων, το οποίο το εξετάζουμε λοιπόν και επίσης εξετάζει το ενδεχόμενο μετασκευής ε, στους μελλοντικούς κανόνες Euro 7, ως έκτο κανόνα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ε, βρισκόμαστε σε προπαρασκευαστικό στάδιο ως προς τη στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος πάλι σε εσά. Σας ευχαριστώ. Να απαντήσω πρώτα στις ερωτήσεις ε, του κυρίου Γκερμπράντη για τον έλεγχο της αγοράς και την εφαρμογή της νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη. Τι γίνεται λοιπόν με τα ελεγκτικά όργανα των ε, κρατών μελών. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους και είναι φυσικά ελεύθερα να επιλέξουν τον τρόπο που θα γίνουν οι έλεγχοι και ποιος θα τους διεξαγεί. Συμφωνούμε όμως μαζί σας και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μαζί τους στην ε, Επιτροπή Επαφής, όπου θα συμμετάσχουν όλοι. Και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να γίνει και μια παρόμοια μελέτη σε εθνικό επίπεδο γιατί και από τις ε, συζητήσεις της ε, περασμένης εβδομάδας και από όσα αναφέρει ο τύπος έχουμε ανταπόκριση πάνω από 95% στη Γερμανία σχετικά με το ενημερωτικό μας έγγραφο. Και είπατε στην τελευταία σε συνεδρίαση ότι ίσως τα κράτη-μέλη δεν είναι αρκετά ενημερωμένα για το θέμα αυτό και θα έπρεπε να εντείνουν τις προσπάθειες τους για επίλυση του ζητήματος. Τώρα η μετασκευή στο υλικό κομμάτι. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφέρει τις προθέσεις της, οπότε δεν νομίζω πως ε, είναι δυνατό να δώσει απάντηση το ηλεκτρικό, ελεκτικό συνέδριο. Είναι δικαιοδοσία των ε, κρατών μελών. Οπότε εμεί δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Volkswagen, ε, είναι ένα ενημερωτικό έγγραφο. Έχουμε δημοσιεύσει αυτό που είναι εφικτό να δημοσιευτεί. Συνεχίζονται οι συζητήσεις, οπότε δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωμοδοτήσουμε για το αν η διαφωνία είναι σωστή ή όχι, διότι δεν γνωρίζουμε πώς έχει εξοδέψει το, τα ποσά αυτά η Volkswagen. Οπότε δεν μπορώ να σας δώσω μία σαφή απάντηση σε αυτό το θέμα. Έτσι έχω λοιπόν καταλάβει τις ερωτήσεις που μας κάνατε. Σας απάντησε και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της μετασκευή, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ε, κύριε Μπράντι, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι. Ε, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζέικοπ για τις απαντήσεις. Ε, έχω μία επιπλέον ερώτηση. Το κυριότερο πρόβλημα είναι τα οχήματα με αυτό το λογισμικό εξαπάτηση και το πρόβλημα επιμένει διότι δεν έχει λυθεί ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπουμε εθνικέ λύσεις όπως ε, της Γερμανίας, όμως δεν υπάρχει ε, κάτι παραπάνω. Πούμε, στη Γερμανία προσφέρουν 6.000 ευρώ για ε, τα πειραγμένα αυτά οχήματα. Ε, τα οχήματα όμως αυτά θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται σε άλλα κρατημέλη γιατί θα γίνουν πιο φτηνά, θα χρησιμοποιηθούν για εξαγωγές. Ένας οργανισμός στην Ευρώπη όμως ε, έχει τη δυνατότητα να συντονίσει την ε, ανταπόκριση αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτός ο οργανισμός είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε όμως ε, έλλειψη ανταπόκρισης. Τι προτίθενται λοιπόν να κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να επιληθεί το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρά να αφήσουν την λύση στα κράτη-μέλη σε κάθε κράτος μέλος από μόνο του με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί σε διοργανικό επίπεδο και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Δεν μπορώ λοιπόν να σας δώσω μία σαφή απάντηση σχετικά με το τι ε, μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς πρώτερη συμφωνία με τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται μια εναρμονισμένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν πρέπει να αφήσουμε το κάθε κράτος μέλος μόνο του. Τώρα, οι εξαγωγές ε, δεν θα γίνουν ενδεχομένως μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε τρίτες χώρες. Σε αν το κοιτάξουμε παγκόσμια το θέμα, σίγουρα με αυτή την προσέγγιση δεν πρόκειται να επιληθεί το πρόβλημα. Στις Ηνωμένε Πολιτείες δεν επιτρέπονται αυτές οι ενδιάμεσες λύσεις ή γίνεται μετασκευή ή πετάς στο αυτοκίνητο. Επίσης, οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα δεν θα γίνουν άμεσα αίσθητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η συνάντησή μας, ε, η πρωινή μας συνεδρίαση. Θα σας δω όλους το απόγευμα.